Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη φτάνουμε στις προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία. Θα ζητήσω από όλους τους ομιλητές να σεβαστούν τον χρόνο αγόρευσής τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Πρώτα απ' όλα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Ιντβελντ εκ των ε, συγγραφέων για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, Επίτροπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε σήμερα νομοθεσία που μπορεί να ψηφιστεί από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο και που ενδεχομένως θα επιδράσει αρνητικότατα στην θέση των διεμφυλικών στη Λιθουανία. Είναι ατυχές το γεγονός ότι το ξανασυζητάμε το θέμα γιατί ήδη έχει ε, ψηφίσει επ' αυτού το Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα που προτείναμε για την αυριανή ψηφοφορία είναι ξεκάθαρο. Απευθύνουμε έκκληση στους Λιθουανούς συναδέλφους να στοχαστούν το θέμα καλύτερα και να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία που θα ψηφίσουν δεν θα οδηγήσει σε διακρίσεις σε βάρος των λεγόμενων διεμφυλικών ατόμων. Δεν νομίζω ότι έχω να πω πολλά για το ψήφισμα καθ' αυτό. Πιστεύω όμως ότι όλο και σαφέστερο γίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξοπλιστεί με ισχυρότερα νομικά εργαλεία για την επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάναμε συζητήσεις για τον αμφιλεγόμενο Ουγγρικό νόμο για τα ΜΜΕ πρόσφατα και αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα. Εμείς έχουμε θεσπίσει αρχές, κοινέ αξίες 500 εκατομμυρίων πολιτών στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Όταν όμως πάμε να τις εφαρμόσουμε στην πράξη αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Γι' αυτό, Επίτροπε, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για την πρότασή μας για έναν ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των διεμφυλικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν έκανε πολλά για την ισότητα των φύλων και έχουμε τους ε, τακτικούς οδικούς χάρτες για την ισότητα των φύλων. Έχουμε πολλές στρατηγικές καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού Έχουμε πολλές στρατηγικές για την ενίσχυση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν έχουμε όμως για τους διεμφυλικούς. Νομίζω ότι είναι κατεπήγον και αναγκαίο να υπάρξει μια τέτοια στρατηγική που θα καταπολεμήσει τις, ε, την άγνοια, της διακρίσεις, ε, της προκαταλήψεις, της διακρίσεις και θα ενισχύσει τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Σήμερα συζητάμε για τις τροπολογίες που κατετέθησαν στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας απομακρύνει από το γεγονός ότι, ότι η ομοφοβία υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτρόπου και να ακούσω τις απόψεις για ένα άλλο θέμα επίσης που αφορά την πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αιτούντες άσυλο που ζητούν άσυλο γιατί διώκονται λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού σε ένα κράτος μέλος που δεν θα το αναφέρω πρέπει να περάσουν από φαλομετρικό τεστ έτσι λέγεται αυτό το πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα εξευτελιστικό δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα και θέλω να ακούσω τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λούνατσεκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφε. Η συνάδελφος κυρία Ιντεβέλτ εξήγησε την, ε, το ψήφιμα και αναφέρθηκε σε αυτό και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ μαζί της και θα ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ σχετικά με τον δικό χάρτη για τα δικαιώματα των ομοφυλοφύλων, αμφιφιλόφιλων και διεμφυλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ωστόσο θα ήθελα να πάρω μια άλλη οπτική γωνία και να πείσω εκείνους στο Κοινοβούλιο που δεν αποφάσισαν ακόμα να υπερψηφίσουν αυτό το ψήφισμα. Γνωρίζετε ότι για τα ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Σοφία Φέλτ, ο Μάικλ Κάνσμαν και εγώ ήδη αντιπροσωπούμε αντιπροσωπεύοντας ομάδα ομάδες του Κοινοβουλίου επισκεφθήκαμε το Βίλνιους στη Λιθουανία όπου θα γινόταν η πρώτη παρέλαση περηφάνεια στο Βίλνους αντιπροσωπεύουν τους ομοφιλόφιλους, ομοφιλόφιλους και διεμφυλικούς στην πόλη αυτή. Και εμείς ε, είμαστε κάτω από, την Ευρωπαϊκή, από τις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας ότι προστατεύει αυτές τις ομάδες ανθρώπων και στη Λιθουανία. Τώρα, ε, τι θα συμβεί σε εμά και στους Λιθουανούς που τον άλλο χρόνο θα συμμετάσχουν σε αυτή την παρέλαση στο Βέλνιος εάν εγκριθεί αυτός ο νόμος. Ε, ξέρετε ότι καθένας από μας ε, θα μπορούσε να πληρώσει ένα πολύ ψηλό πρόστιμο ε, για την λόγω δημόσιας προβολής ομο, της ομοφιλοφιλίας, ομοφιλοφιλικών σχέσεων, παραδείγματι. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια χώρα που πάλεψε για την, δική της, για την ελευθερία της πριν από 20 χρόνια και όπου και οι ομοφιλόφιλοι και αμφιφιλόφιλοι και αυτοί υπάλεψαν για την ανεξαρτησία της Λιθουανίας. Ο πρόεδρος της ε, Λιθουανίας ε, και η κυβέρνηση είπαν ότι αυτός ο νόμος αντιβαίνει το σύνταγμα της Λιθανίας και ελπίζω ότι θα καταστήσει σαφές ότι οι διαφορετικές μορφές έκφρασης σεξουαλικού προσανατολισμού ή μορφές διαβίωσης αποτέλεσαν τμήμα όλων των πολιτισμών και όλων των κοινωνιών και στη Λιθουανία. Ε, και ε, το να ε, συγκαλύπτει κανείς τα πράγματα στους νέους ανθρώπους με τον τρόπο αυτό ενισχύει ε, φαινόμενα μυσαλλοδοξίας και μίσους. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα ήθελε κανείς μας για την Λιθουανία. Ελπίζω λοιπόν ότι εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επισφίσετε το ψήφισμα. Τη δική σας υποστήριξη πιστεύω ότι την έχουμε ούτως ή άλλως. De Jong, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι δύο προλαλήσασε συνάδελφοι, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Μια, ένα άλλο, μια άλλη πλευρά της προβληματικής. Βεβαίως αυτή η τροπολογία ε, στον διοικητικό κώδικα ε, της Λιθουανίας ε, μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη Λιθουανία. Αλλά μπορεί να θεωρηθεί και σαν παράδειγμα αναφοράς και σε άλλους όπου αναγνωρίζονται οι ενώσεις των ομοφιλοφίλων σε άλλες χώρες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ε, θα ήθελα να μάθω εάν η Λιθουανία ε, θα δεχτεί ε, ζευγάρια από κατηγορίες ΛΟΑΔ για περιπτώσεις ζευγαριών που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, η αναγνώριση του δικαιώματός τους ε, είναι πλέον από πέρσι δεδομένη. Επίσης, ε, θα ήθελα να ξέρω εάν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκαναν κάποια ανάλυση για την αναγνώριση ενώσεων μεταξύ μελών ε, ΛΟΑΔ. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ρουμανία πούμε, που δεν δέχτηκαν τέτοιου είδους ε, ζευγάρια. Ε, πρόσφατα παρουσιάστηκε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μία έκθεση σχετικά με την ομοφοβία ε, γνωρίζουμε λοιπόν ότι σε πολλές ε, χώρες της Ευρώπης ε, υπάρχουν προβλήματα, αλλά στη Λιθουανία πραγματικά η κατάσταση είναι έκτακτη και χρειάζεται οπωσδήποτε άμεση απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα για δύο λεπτά. Καλησπέρα σας, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να πω ειλικρινά ότι αδυνατό να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει στη Λιθουανία. Ε, τώρα που βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε κάνει μια πρόοδο σχέση με το τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τώρα οι χώρες μέλη αποστέλουν μηνύματα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ε, θεωρούμε ότι η θέσπιση ενός τέτοιου νόμου είναι τελείως οπισθοδρομική και αγνοεί το τι έχουμε πετύχει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα η προστασία των νέων ανθρώπων υπό την έννοια αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πρόσχημα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους έναντι φτώχειας, βίας και πρέπει να εξασφαλίσουμε κατάλληλες προϋποθέσεις εκπαίδευσης και σωστής ανάπτυξης. Αλλά όλοι μας γνωρίζουμε από την ιδία μας πείρα ότι τα παιδιά δεν ενοχλούνται από την έκφραση αγάπης άλλων ε, μορφών ε, έρωτα πλην του ετεροφιλοφιλικού. Ε, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε υπό ποια έννοια η θέση αυτή είναι εσφαλμένη. Ο νόμος στην Λιθανία είναι εσφαλμένος. Ε, και παραβιάζει, αντιβαίνει στις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, δεν σέβονται το δικαίωμα έκφρασης, ε, το δικαίωμα του συνέρχεσης και την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού. Κύριε Πίτροπε, θα Εάν ο νόμος εφαρμοστεί, ε, πρόκειται η Επιτροπή να κινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση κατά της Λιθουανίας. Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Because καταδικάζει ε, την ε, ομοφοβία και κάθε μορφή της. Ε, και άλλωστε την 22 Νοεμβρίου 2010 επισκέφθηκα τη Λιθουανία και συζήτησα με τον πρόεδρο της χώρας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αυτήν την τροπολογία στο Διοικητικό Κώδικα που δημιουργεί νέο αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο για, παραθέτω, δημόσια προβολή ομοφιλοφιλικών ε, σχέσεων σε ε, δημόσιους χώρους καθώς επίσης ε, και μία πρόταση για αντίστοιχη τροπολογία και τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Πρέπει να σας πω ότι δύο φορές αναβλήθηκε η ψηφοφορία της τροπολογίας αυτής στο Διοικητικό Κώδικα ε, και τώρα θα λάβει χώρα η νέα ψηφοφορία τον, ε, την Άνοιξη. Ε, γίνεται, μελετάτε το ενδεχόμενο τροποποίησης του διοικητικού κώδικα, του ποινικού κώδικα και άλλων νόμων της Λιθωανίας υπό το φως του σεβασμού των, και της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από καιρό έχει εκφράσει ε, την, ε, ε, το, τους ενδιασμούς της όσον αφορά την τροπολογία αυτή, κυρίως δε σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων και σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων. Το Δεκέμβριο του 2009 τροποποιήθηκε για μία ακόμα φορά ο, ο νόμος αυτός και αφορούν και αφορά πλέον ε, ε, τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να προβάλλουν σεξουαλικές σχέσεις ή ορισμούς του γάμου ή των συστατικών στοιχείων μιας οικογένειας διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται στο Σύνταγμα ή στον αστικό ε, κώδικα και ε, αυτό με το σκεπτικό ότι μπορούν τέτοιου είδους, ε, ε, τέτοιου παραδείγματα να δημιουργήσουν πρόβλημα στα, στους ανηλίκους. Αλλά βεβαίως με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερης πληροφόρησης καθώς επίσης και της, του σεβασμού των ελευθεριών, των προσωπικών ελευθεριών. Όσον αφορά τώρα την ε, παροχή πληροφοριών, ε, νόμου που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2010, ε, σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε οποιαδήποτε διαφήμιση ή προβολή σε δημόσιο χώρο δεν θα πρέπει ε, να επιδεικνύει, ε, ε, να περιέχει επίδειξη ή προβολή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αλλά και στην περίπτωση αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση με, την, με το άρθρο 21 της, της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και με την οδηγία για την την ε, ε, τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δι, ε, αντέδρασε στην ακύρωση τελευταία στιγμής της, της πορείας υπερηφάνειας της Gay Pride Parade και θεώρησε ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 12 ε, της ε, χάρτας καθώς επίσης ε, και των βασικών αρχών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήδη την 8η Μαΐου του 2010 προχώρησε σε παρατήρηση κατά της Λιθουανίας. Τώρα, την, το, η δυνατή Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της ομοφοβίας. Κατά αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι η προτεραιότητα είναι η πλήρη συμμόρφωση των νομοθεσιών ε, με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ε, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 21 της ίδιας χάρτας. Πώς μπορεί να γίνει η συμμόρφωση αυτή. Αυτό εξηγήθηκε σαφέστατα στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, για την στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έτσι όπως εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και βεβαίως θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό ε, στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που καλύπτει βεβαίως και την ε, πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 20 αυτό θα γίνει την άνοιξη του 2011. The phallometric. Κατά αυτή την έννοια, ε, αυτές οι φαλομετρικές ε, ε, μετρήσεις στη διαδικασία ασύλου ενσωματώνεται ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και άρα σχετίζεται άμεσα με το άρθρο 21 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 21 απαγορεύει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και αναφέρει σαφώς ότι εάν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έτσι όπως εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο ε, ε, υπάρχει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση τότε ε, υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Επομένω, είναι σαφ, καθίσταται σαφέ ότι έχει δικαίωμα και δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να επαναλάβω την ε, σαφή ε, ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση οποιασδήποτε εκδήλωσης ομοφοβίας. Όσον αφορά τώρα την αναγνώριση του, της οικογενειακής κατάστασης. Δεν προτιθέμεθα να προτείνουμε οποιαδήποτε νομοθεσία η οποία θα παρεμβαίνει ε, στο ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών ή που θα μπορούσε να τροποποιήσει τον εθνικό ορισμό του γάμου. Αυτό ε, αφορά την επικουρικότητα. Αμοιβαία αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης ε, αφορά τις δύο συνοριακές σχέσεις όπως ας πούμε το, τα πιστοποιητικά γέννησης και δεν αφορούν τον γάμο. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε λοιπόν τα πράγματα. Τα εθνικά κράτη είναι αυτά τα οποία ορίζουν τι σημαίνει γάμος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία και την άρση οποιασδήποτε πρακτικής μεταχείρισης. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξέρουμε τι προβλέπει ε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και μόνο τα προβλεπόμενα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο εις τους αγορητές εξ των πολιτικών ομάδων. Ξεκινούμε με τον κύριο Μπουζούτιλ, δύο λεπτά για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΛΚ έχει δεσμευτεί να και αρχές της Ένωσης, ιδιαίτερα τα θερμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει η Ευρώπη να καταπολεμήσει κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Παράλληλα πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα κάθε δημοκρατίας στο βαθμό που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή των μη, της μη διάκρισης για να συζητούμε, να τροποποιούμε και να εγκρίνουμε εθνική νομοθεσία χωρίς να παρεμβαίνουμε στην αντιπαράθεση στα εθνικά κοινοβούλια χωρίς να παραβιάζουμε την αρχή της επικουρικότητας και χωρίς να καταδικάζουμε προώρα ένα κράτος μέλος. Δεν μας αρέσει η ιδέα της καταδίκης ενός κράτους μέλους, ιδιαίτερα επειδή εν προκειμένου η προτινόμενη τροποποίηση ακόμα δεν έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Λιθουανικού Κοινοβουλίου και ακόμα είναι υπό αναθεώρηση από τις λιθουανικές αρχές. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις επίσης έχουν θεωρηθεί ότι αντιβαίνουν ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τις ίδιες λιθουανικές αρχές που εδήλωσαν ότι θα αναλάβουν δράση για να διορθωθεί η κατάσταση και να τύχει σεβασμού η αρχή των μη διακρίσεων βάση γενετήσιου προσανατολισμού. Η προτινόμενη λοιπόν νομοθεσία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα φτάσει να γίνει καταστατικός νόμος της Λουθουανίας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να καταδικάσουμε πρόωρα τη χώρα αυτή, τη χώρα μέλος. Τέλος, ε, ελπίζω παρόλα αυτά ότι αύριο το ΕΛΚ θα μπορέσει να υποστηρίξει το κοινό ψήφισμα στο βαθμό που δεν καταδικάζει κάποιο μεμονωμένο κράτος μέλος και στο βαθμό που θα τροποποιηθεί ώστε να έχει μεγαλύτερη ισορροπία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριο Μωράη απουσιάζει, Επομένω, θα δώσω αμέσω τον λόγο εξ ονόματο των ε, ελευθέρων στην κυρία Λάτφορντ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι η Λιθάνια θα διδαχθεί από την εμπειρία τη μεγάλη Βρετανία, η οποία είχε τα δικά τη ε, προβλήματα ε, σχέση ένα νόμο ο οποίο απαγόρευε την ε, προβολή της σεξουαλικότητας στα σχολεία. Το... Ο Ντέιβιτ Cameron είπε ότι πριν από 18 μήνες το κόμμα του έσφαλε υποστηρίζοντας αυτό το νόμο του 98 ο οποίος ε, τώρα καταργήθηκε. Ο Ντέβιτ Κάμερον ε, είπε ότι ο πρώτος γκέι υπουργό στη Μεγάλη Βρετανία θα είναι ένας ε, τόρι. Αυτή η εξέλιξη στις ε, ε, νοοτροπίες αντανακλάται σε ένα μάλλον αρκετά ήπιο ψήφισμα. Ε, ελπίζω ότι το ΕΛΚ θα μπορέσει να προσυπογράψει το ψήφισμα αυτό εάν τα περισσότερα μέλη της το στηρίξουν. Ε, η διοκτησία ε, ενός πανδοχείου στη Μεγάλη Βρετανία υποχρεώθηκαν να πληρώσουν αποζημίωση σε ένα γκέι ζεύγος το οποίο αρνήθηκαν τη διαμονή εκεί. Ε, είναι δυνατόν να συζητηθούν οι απόψεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε σχέση με τις ε, ομοφυλόφιλες σχέσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζονται διακρίσεις εις βάρος ομοφυλοφίλων το να απαγορεύεται η πρόθεση των σχέσεων αυτών έχει μια δυσμενή επίδραση στη δημόσια, στην ελευθερία του λόγου. Ε, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους στις, ε, όλες τις πολιτικές ομάδες ε, σε αυτό το σώμα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τους πρασίνους, Κορνέλισεν, για ένα λεπτό. Η κυρία Κορνέλισεν. Κυρία. Πρόεδρε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στην Λιθουανία ε, παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Οι αξίες και οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές αλλά κάρτε όποια χώρα θέλει να γίνει μέλος και να παραμείνει μέλος θα πρέπει να σέβεται όλες τις χώρες. Αυτό ισχύει για τη Λιθουανία αλλά και την Γαλλία και τις ε, κάτω χώρες ε, στην περίπτωση που επιθυμούν η κάτω χώρες να συρρυκνώσει τα δικαιώματα των ε, προσφύγων ή των μεταναστών. Χαίρομαι που ο Επίτροπος ε, ζήτησε να διεξαχθεί μια νομική ανάλυση και θα λάβει περαιτέρω βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να γίνονται θύματα μιας τέτοιας νομοθεσίας και ε, κατ' ουσία να ζητούν την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περιπτώσεις παραβιάσεων. Ο κύριος Τάνοκ, για δύο λεπτά. Η βασική αρχή είναι τα ίσα δικαιώματα και ελευθερίες. Η βασική αρχή της Ένωσης και τα κράτη-μέλη και τα ενδεχόμενα κράτη-μέλη θα πρέπει να σπαστούν τις αρχές αυτές και τον χάρτη των δικαιωμάτων. Όταν πριν από 7 χρόνια έγινε μέλος η Λιθουανία, σπάστηκε τις αρχές αυτές της ανεκτικότητας. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, άρθρα 12 και 21, τέθηκαν σε ισχύ και έδωσαν κι άλλες ε, διασφαλίσεις στους ανθρώπους με διαφορετικό από τον της σεξουαλικό προσανατολισμό. Κατηγορηματικά λέω ότι η ομάδα μου ε, είναι υπέρ των αρχών της ανεκτικότητας παντού πολύ. Ευρωπαίοι όμως είναι παραδοσιακοί σε ό,τι αφορά την ε, ομοφιλοφιλία ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει νόμος και για τους ΛΟΑΔ, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ευκαιρία να εκφραστούν διαφορετικές, όχι εμπριστικές βέβαια, απόψεις. Και εκείνοι πρέπει να είναι ελεύθερη. Σίγουρα η λιθουανική κοινωνία παραμένει πολύ συντηρητική. Πρέπει να το καταλάβουμε είναι, δικαιούνται να έχουν τις απόψεις τους. Αλλά σε νομικό και θεσμικό επίπεδο δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε την αρχή της ισότητας που είναι το χαρακτηριστικό της των προοδευτικών κοινωνιών της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν και τα ατομικά δικαιώματα να διασφαλίζονται και αυτό πραγματικά έδρασε ως μαγνήτης στους Λιθουανούς μετά τον κομμουνισμό. Απευθύνω έκκληση στις Λιθουανικές αρχές να σκεφτούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να προλαμβάνει την περιθωριοποίηση, τη δίωξη ε, μειονοτήτων που ήταν τόσο συνήθισε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε το νομοθέτημα στην εξέλιξή του και να δούμε αν το νομοθέτημα αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο κύριος Μπουσουτήλ ε, είπε ότι είναι πολύ πιθανό το νομοσχέδιο να μην γίνει νόμος. Η Λιθουανία είναι δημοκρατία και γνωρίζει πολύ καλά τα τεράστια ζητήματα που θα προκύψουν αν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Ενωτική Αριστερά τώρα και ο κύριος Χίγκινς για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, το προτινόμενο ε, νομοθέτημα για την ε, παρεμπόδιση ομοφιλοφιλικών σχέσεων και διαφημίσεων ε, αποτελεί απειλή για όλους τους ΛΟΑΔ. Είναι τραγικά ηρωνικό το γεγονός ότι μια χώρα που φόρεσε τις χειροπέδες του σταλινισμού και αυτό πριν από 20 χρόνια τώρα ε, πισωγυρίζει σε ένα από τα δικήματα εκείνου του καθεστώτος. Δηλαδή ε, την ανεκτικότητα απέναντι σε ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ε, ε ήταν ε, δυσάρεστη και πραγματικά είναι απογοητευτικό να παρεμποδίζεται η πορεία της περηφάνειας ή να ε, δημιουργούνται από διοπομπέοι τράγοι. Ε, ο καπιταλισμός, η να δημιουργουνται απο δυο πομπει έχει καταστρέψει τις βαλτικές δημοκρατίες και τη Λιθουανία όπου η ανεργία των νέων έφτασε στα 45% και γενικά 18%. Είναι κοινικό τρόπος να παρακάμπτεται ε, έτσι η προσοχή από τα βασικά. Η εκστρατεία ομοφοβίας ε, στηρίζεται στο ότι ε, δημιουργούνται απειλές για τους νέους. Αυτό είναι παραπλανητικό, είναι δυσφήμιση, είναι συκοφαντία. Ε, είναι λάθος οι γονείς να πάνε έτσι να προστατέψουν τα παιδιά τους στην ε, Αγγλία ε, υπήρχαν ε, περιοχές υπεράνω υποψίας όπως η Καθολική Εκκλησία και όμως είδαμε τι συνέβη. Είναι δύσκολο πολλές φορές να αντιμετωπιστεί η παιδική σεξουαλικότητα. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς φόβο, με ανεκτικότητα. Στη Λιθουανία, στη Ρωσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού οι άνθρωποι θα πρέπει να ζουν ειρηνικά και σύμφωνα με την ταυτότητα που έχει ο καθένας τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συμπράσας νομίζω δεν είναι στην αίθουσα. Ε, περνάμε στους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος ε, Στογιάννοφ, 1,5 λεπτό. Κυρία Επίτροπε. Που κύριε Επίτροπε, η κατάσταση αυτή μου θυμίζει μια ταινία όπου η τοπική αστυνομία καταδίκασε τους ανθρώπους πριν από τα εγκλήματά τους βασιζόμενοι σε αυθαιρεσίες. Βλέπουμε και εδώ ότι ο λιθωνικός ε, λαός καταδικάζεται για κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει. Ε, Πρόκειται εδώ για μια σύγκρουση μεταξύ ε, νομοθεσιών μεταξύ διαφόρων χωρών και διαφόρων ομάδων. Μιλούμε για το δικαίωμα του συνέχεια, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ευσταθεί. Ε, μιλούμε για μια ειρηνική συνάθρηση ορισμένων ανθρώπων που δεν παραβιάζει τον νόμο. Και νομίζω ότι μελλοντικά θα υπάρξει μια σύγκρουση δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να κρίνουμε ε, ποια δικαιώματα ε, ε, προηγούνται έναντι άλλων εάν εξετάσουμε ακριβώς μια τέτοια επέκταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι. Ξεκινάμε με την κυρία Σκριντλεύσκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή στην Λιθουανία η κατάσταση είναι τέτοια όπου από την μία πλευρά η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση μπορεί να νομοθετήσει ελεύθερα, από την άλλη πλευρά όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται από, τον, από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ε, τις ε, διεθνείς συνθήκες. Επομένως πρέπει να επαγρυπνούμε για περιπτώσεις παραβίασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και αν πρόκειται για τον γενετήσιο προσανατολισμό των ατόμων. Πρόκειται για παραβίαση των δικαιωμάτων του ε, τόμου και ενδεχομένως η τροπολογία του διοικητικού κώδικα ενδεχομένως θα μειώσει την ελευθερία έκφρασης ε, λόγω του γενετήσου προσανατολισμού. Γι' αυτό λοιπόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς προσπαθήσαμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εθνικές μειονότητες στην ε, Λιθουανία γιατί δεν τους δίδονται τα ίδια δικαιώματα ούτε χαίρουν του ιδίου σεβασμού με τους υπόλοιπους ε, πολίτες. Πρέπει να δημιουργηθούν, ε, πρέπει να γίνουν ειδικέ αναφορές στην κοινωτική νομοθεσία και να περιλαμβάνονται και οι εθνικές μειονότητες. Ευχαριστώ πολύ. Μπλίνκε Βυσιούτε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή συζητούμε ένα θέμα που είναι ευαίσθητο για τη χώρα μου. Και θέλω εξ αρχής να πω ότι όσα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Λιθουανία σέβεται ε, τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι ατυχές που κάποιοι μεμονωμένοι βουλευτές ε, του Λιθουανικού Κοινοβουλίου ξεκίνησαν ε, κάποιες τροπολογίες οι οποίες αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα βεβαίως η συζήτηση της τροπολογίας. Πάντως σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτή η τιμωρία με πρόστιμα για δημόσια προβολή σχέσεων και απόψεων, οπωσδήποτε αυτό θα αποτελεί διακριτική μεταχείριση ε, βάσει, του γενετήσιου προσανατολισμού και θα αποτελεί παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, και τη Νομοθεσία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για, έναν, ε, για μια τροπολογία η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή ακόμα και έχει μάλιστα ε, ε, έχει μάλιστα αποτελέσει αντικείμενο ε, άρνησης από πλευράς του Προέδρου της Λιθουανίας. Είναι γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια διεθνής επίκριση όσον αφορά το ζήτημα αυτό και το Λιθουανικό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι τελικά θα καταψηφίσει την τροπολογία αυτή που δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος ε, Ρωμέβα η Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ε, κατέστη σαφές μήνυμα προς το Λιθουανικό Κοινοβούλιο, αλλά όχι μονάχα σε αυτούς, όλους, προς όλους αυτούς που εξακολουθούν να συζητούν πολύ βασικά ζητήματα. Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε κάποιους συναδέλφους που φαίνεται ότι τα λησμονούν. Το ένα είναι ότι η ομοφιλοφιλία δεν ε, θεωρείται πλέον ασθένεια. Και το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη έρευνα που να καταδεικνύει ότι η ε, διαπαιδαγώγηση, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μπορεί να δημιουργήσει ότι μπορεί να επηρεάσει λοιπόν την, ε, το σεξουαλικό του ε, προσανατολισμό. Ε, Επομένω, θεωρώ ότι είναι αστείο ακόμα και το να συζητούμε τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει το ψήφισμα και θα πρέπει να στηρίξουμε τον πρόεδρο τη Λιθουανία στην προσπάθειά του να σταματήσει τη συζήτηση αυτή. Αλλά αυτό δεν ισχύει μονάχα την Λιθουανία. Ισχύει για όλου αυτού που εξακολουθούν να θέλουν να συζητούν αυτού του είδου τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Σιμάνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει πιο ευαίσθητο κοινοβούλιο όταν πρόκειται για την προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού από το ευρωπαϊκό. Το λιθουανικό νομοσχέδιο ηρωνικώς μεταφράστηκε και καταδικάστηκε προτού καν εγκριθεί. Δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στην ε, κυρίαρχη νομοθετική διαδικασία ενός κράτους μέλους. Θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην νομοθετική διαδικασία στη Λιθουανία. Πρέπει να δείξουμε περισσότερη κατανόηση προς τους Λιθουανούς εθνικούς βουλευτές οι οποίοι φροντίζουν να προστατέψουν τα παιδιά απέναντι σε επιθέσεις σεξουαλικού περιεχομένου. Τα παιδιά δεν τα λαμβάνετε υπόψη στη συζήτησή σας καθόλου. Ούτε επιδεικνύεται σεβασμό στην, ε, στα κυρίαρχα δικαιώματα ούτε σκέφτεστε τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το κείμενο αυτό, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Μια και αποσιάζει ο Σλάνθος Χέντε, θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Σενίζιν για ένα λεπτό. Στην κυρία Ζενίση. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι επισμένοι για την ισότητα των δικαιωμάτων τους, αλλά σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το επίπεδο της ανεκτικότητας προς ε, σεξουαλικές μειονότητες ε, είναι μειωμένο. Υπάρχουν περιπτώσεις επιθετικότητας κατά των μειονοτήτων αυτών, ε, απαγορεύσεις των ποριών τους και νομοσχέδια όπως αυτό τώρα στη Λιθουανία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει το ίδιο ελάχιστο επίπεδο προστασίας κατά των διακρίσεων λόγω του, των, της αναπηρίας του σεξουαλικού προσανατολισμού, του AIDS ή κάποιων πεπιθήσεων. Πρέπει λοιπόν να γίνει, υπάρξει και διαχωρισμός κράτους εκκλησίας γιατί η ομοφοβία υπάρχει ιδιαίτερα εκεί όπου η θρησκεία, η εκκλησία παίζει σημαντικό ρόλο και πολύ ισχυρό. Στα Ισλαμικά κράτη για παράδειγμα η ομοφιλοφιλοφιλία τιμωρείται με ποινή θανάτου. Πρέπει λοιπόν να προασπίσουμε την ελευθερία και το ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τροτμάνα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η τροποποίηση σε σχέση με την δημόσια προβολή της ομοφιλοφιλίας διατυπώθηκε στο πλαίσιο του νόμου για την προστασία των αναλύκων ε, κατά των επιζήμιων συνεπειών της δημόσιας ενημέρωσης. Πώς είναι δυνατόν να θέλει κανείς ε, να προσπίσει τα δικαιώματα των ανηλίκων ε, παραβιάζοντας το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Όλοι εδώ γνωρίζουμε ότι ένα τέτοιο κείμενο επιφέρει την συγκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού και επανέρχεται οπισθοχωρή εναντί κάποιων δικαιωμάτων τα οποία έχει υπερασπιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταυτόχρονα σε μια συγκυρία όπου γινόμαστε μάρτυρες επιθετικών πράξεων κατά των ομοφιλοφίλων. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια παρότρινση προς την κατεύθυνση της ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας ή πρόκειται για μια έκκληση, ένα κύμα ε, βία, ε, ενίσχυσης της βίας. Ε, οδηγούμεθα λοιπόν σε μια κλειστή κοινωνία η οποία δεν λαμβάνει υπόψη το σεβασμό έναντι των δικαιωμάτων των άλλων. Και αυτό αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές αξίες που διακινούνται ακριβώς από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διαφύλαξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών ελευθερων ελευθεριών. Επίσης αντιβαίνει ε, σε όλο το κόρπους της ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση των ε, διακρίσεων και ενώ επιθυμούμε ε, περισσότερη ισότητα εντός των κοινωνιών μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπη που εδώ εκφράσατε πολύ ξεκάθαρες απόψεις και θα ήθελα όλες οι πολιτικές ομάδες να εισακούσουν τα επιχειρήματά σας καθώς και αυτά των συναδέλφων μου και θα ήθελα να σας πω ε, πόσο ε, επιθυμώ να παρατρύνω τους συναδέλφους όλων των πολιτικών ομάδων να υπερψηφίσουν αυτό το ψήφισμα και να συγχαρώ τους συντάκτες αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Για μία ακόμα φορά σας παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο εργασίας σας, γιατί στις 12 ακριβώς πρέπει να σταματήσουμε. Η κυρία Ζαμπόσκα είναι πρώτη γραμμένη στη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί συζητά το Κοινοβούλιο την τροπολογία που υπέβαλε ένας ε, ε, βουλευτής μίας ενός κοινοβουλίου και ακόμα δεν έχει γίνει νόμος του κράτους. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τι συζητούμε και τι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δηλαδή αύριο, ε, σήμερα κάνουμε μια συζήτηση και αύριο θα γίνει μια ψηφοφορία για μια τροπολογία η οποία δεν έχει ψηφιστεί, η οποία δεν έχει γίνει νόμος και η οποία αφορά απλώς μια συζήτηση που ακόμα γίνεται, λαμβάνει χώρα ε, στην ε, Λιθουανία. Έχουμε την ίδια αίσθηση και για την ε, τροπολογία της Ουγγρικής κυβέρνησης όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Ε, ενώ είπαμε ότι θα αφήσουμε την διαδικασία ε, να ολοκληρωθεί, τελικά συζητούμε για πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν περάσει. Μιλάμε εδώ για κάτι που δεν έχει γίνει αποδεκτό από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο. Παρόλα, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι Λιθουανή. Μιλούμε για ένα ψήφισμα απόψε που στηρίζεται σε μια τροπολογία του διοικητικού κώδικα. Η νομοθετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρεί να παρέμβει. Δεν έγιναν συζητήσει στην Επιτροπή. Σημειώνω δε ότι υπήρξαν και γνωμοδοτήσεις αρνητικές στο νομοσχέδιο. Δεν στηρίζω το ψήφισμα γιατί αποτελεί υπερβολική αντίδραση. Θέλω επίσης να αναφερθώ στον συνάδελφο Χίγκινς και να του πω να μην μιλάει για πράγματα που δεν έχει ζήσει και δεν θα πρέπει να συγκρίνει την, Σοβιετική, την πρώην Σοβιετική Ένωση με τη Λιθουανία. Αυτό είναι κατανόητο για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σταΐν. Η κυρία Σταΐν. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύουν τη διάκριση βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού. Τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλων των χωρών μελών δεσμεύονται, είναι υποχρεωμένα να καταπολεμούν τι διακρίσει βάσει του γενετησίου προσανατολισμού, βάσει τη συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και του άρθρου 19 για τον τρόπο λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λιθουανία είναι χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δεσμευθεί να αυτές τις, να συμμερίζεται αυτέ τι κοινέ αξίε των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζω το γεγονό ότι η Λιθουανία μετά από το πρώτο ψήφισμα του 2001 ε, δεν έχει εφαρμόσει το νόμο αυτό ε, καθώς και δεν ε, εφαρμόστηκε πρόταση για απαγόρευση της ε, παρέλασης ε, των ομοφιλοφίλων. Όσον αφορά τώρα την επιβολή ε, προστήμου ε, για τη δημόσια προβολή αμοφιλοφιλικών ε, σχέσεων, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της ομοφοβίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ για την παρουσία της εδώ στην Ολομέλεια που σε τόσο προχωρημένη ώρα τονίζει την σημασία αυτού του ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ. Κυρία Πρόεδρε, σημείωσα μεγάλη συμφωνία στο κοινοβούλιο αυτό μεταξύ όλων των μεγάλων πολιτικών κομμάτων επί της αρχής των μη διακρίσεων και πιστεύω ότι αν υπάρξει ψήφισμα που θα αναδεικνύει την αρχή αυτή και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο που αποτελεί υποχρέωση των εθνικών κρατών απέναντι στους κανόνες της Ευρώπης που έχουν προσυπογράψει, νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια σημαντική στιγμή. Οι βουλευτές εκείνοι που είπαν σαφώς ότι εδώ μιλάμε για ένα νόμο που δεν είναι ακόμα νόμος, αλλά μια πρόταση ορισμένων βουλευτών, σωστά κάνουν και το υπογραμμίζουν αυτό, αλλά Θέλω να υπενθυμίσω επίσης εδώ ότι και η πρόεδρος της Λιθουανίας και η κυβέρνηση της Λιθουανίας ξεκάθαρα εκφράστηκαν κατά των προτάσεων αυτών ορισμένων βουλευτών. Ελπίζω ότι ομόφωνα σχεδόν θα καταλήξει η συζήτηση επί ε, αρχών που έχουν ελεύθερα συμφωνήσει τα 27 κράτη-μέλη, αρχές δηλαδή των ευρωπαϊκών οδηγιών μας που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι στις ε, αυριανές συζητήσεις και στην ψηφοφορία θα αναδειχθεί αυτή η στεναρή θέση του Κοινοβουλίου. Ε, το ελπίζω ειλικρινά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπο. Πρέπει να σας πω ότι έχω ε, λάβει δύο ψηφίσματα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, η οποία κλείνει εδώ. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12.30. Η επόμενη συνεδρίαση